για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία για ε, Μικροδιαφορών και Διαδικασία Έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Προμής. Ε, the goes... Το λόγο τον έχει η κυρία Γκέριγκερ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή αυτή, διότι θα ψηφίσουμε την έκθεσή μου, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Περνάει δηλαδή ε, από τρεις προεδρίες του Συμβουλίου Έχουμε συζητήσει εκτενώς ε, την ε, έκθεσή μου, όπως επίσης και τις αλλαγές που έχουν υποβληθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συγητές, όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Πολλές από αυτές τις τροπολογίες εμπλούτησαν το περιεχόμενο του κειμένου μου και το απλούστευσαν επίσης. όπως λέει και το όνομα και ο τίτλος μιλάμε για μικροδιαφορές. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο όρος έθεσε πολλά προβλήματα διότι το μικροδιαφορές ε, σημαίνει πολλά πράγματα σε διαφορετικές χώρες. Πάντως η πλειοψηφία των συναδέλφων δέχτηκαν το όνομα αυτό ε, και, το καθα... και ξεκαθαρίζουμε ότι μιλάμε για διαφορές που φτάνουν το ποσό των 10.000 ευρώ. Πάντως ελπίζω ότι ε, πρέπει να σεβαστούμε τα όσα έχουν γίνει, διότι τελείως δεν έχει κανένα νόημα. Ε, μπορούμε νομίζω να περάσουμε στην ψηφοφορία και να ψηφίσουμε ακριβώς όπως έχουμε αποφασίσει. Ξεκινάμε την ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η τροπολογία. Υιοθετείται η τροπολογία, εγκρίνεται. Τροπολογία 88, υπέρ κατά αποχές καλό θα είναι να κάνουμε μια επιβεβαίωση άρχεται η ψηφοφορία We voting op option one. Ψηφίζουμε την εναλλακτική λύση 1, την option 1. Πέρα της ψηφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. 88. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά αποχέ, αποχές εγκρίνεται. Τριάντα τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της Απορρίπτεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Είμαστε στην τροπολογία υπαριθμών 6. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενενήντα ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. Ωραία, ελέγχουμε το 63. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Σαφέστατα έχει απορριφθεί. 67. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά το ελέγξουμε Γιατί την 67. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπέρ για την 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές. Κάς το ελέγξουμε όμως καλύτερα. Εδώ για την 75, ηλεκτρονική εξακρίβωση. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Ναι, απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπορούμε να το ελέγξουμε βέβαια είμαστε στο 81 στην τροπολογία 81 Πέρα της ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. «82 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά καλό θα είναι να το τσεκάρουμε για την 12. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ογδόντα τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε.

κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά καλό θα είναι να το τσεκάρουμε ναι όντως απορρίφθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να εξακριβώσουμε και για την ε, τροπολογία 1 Όντως απορρίφθηκε. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 27 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα ε, ψηφίζουμε το σύνολο της, ε, του σχεδίου της έκθεσης υπέρ, κατά όχι οφείλουμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της, ε, της έκθεσης του σχεδίου έκθεσης Ψήφισαν όλοι και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Επίσης ε, το ψήφισμα, το νομοθετικό ψήφισμα θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. it been εγκρίθηκε απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ηλεκτρονικά πάλι ψηφίζουμε και ένας ακόμα δεν έχει ψηφίσει εγκρίνεται να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Και περνάμε στην ψηφοφορία για την, ε, για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, TTIP. Ο κύριος Βος είναι ο εισηγητής, που έχει και το λόγο. Ähm, zunächst ähm, möchte ich mich einmal ganz kurz entschuldigen. Καταρχάς να ζητήσω σύντομα συγγνώμη για όλη αυτή τη διαδικασία που έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες, όμως πρέπει ξεκάθαρα να το πω ότι δεν έγιναν τα πράγματα με το βέλτιστο τρόπο. Και αυτό ε, έγινε λόγω του Πάσχα και της ε, επόμενης εβδομάδας. Ε, γενικά δεν μπορέσαμε να έχουμε την κατάλληλη συμμετοχή και να έχουμε όλη την εκπροσώπηση που θέλαμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν και με το τηλέφωνο να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς ε, λόγω των διαφόρων θέσεων ε, που υπήρξαν, όμως ε, δεν ήταν αυτό δυνατό τελικά και γι' αυτό θεωρώ προσωπικά που, ότι είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα ήταν προοδευτικό. Όμως τα πράγματα είναι όπως είναι και γι' αυτό ε, θα ήθελα άλλη μια φορά να μιλήσω ε, και να πω ότι η διαδικασία δεν ήταν η βέλτιστη γιατί χθες μέχρι και αργά το βράδυ έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ζητώ συγγνώμη, ελπίζω να μην επαναληφθεί αυτό όπως και να έχει. Η κυρία Ρέκνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με τον προηγούμενο ε, ομιλητή. Είναι μια καυτή πατάτα η συμφωνία TTIP. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ε, θέσεις που πρέπει να συγκεραστούν ε, για να υπερασπιστώ τον Αντρές να πω ότι η λίστα ψηφοφοριών ήρθε πάρα πολύ αργά. Έχουμε αυτή την συμφωνία κυρίων ε, που ε, λέει ότι πρέπει η λίστα αυτή να είναι στα χέρια μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Ε, συνήθως αυτό συμβαίνει και όταν υπάρχει πρόβλημα πραγματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να το κάνουμε, γιατί εντάξει μέσα σε μια νύχτα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά, όμως ε, δεν θέλω εμείς και η ομάδα μας ε, να πρέπει να ε, ξεφύγουμε από αυτό που έχουμε ήδη αποφασίσει. Και να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία για το γεγονός ότι μπορέσαμε να εργαστούμε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τώρα που ψηφίζουμε να πούμε ότι ένα κομμάτι της λίστας ψηφοφοριών ε, στην ε, τροπολογία 9 συγκεκριμένα βλέπω ότι δεν είναι συμβατό αυτό που λέει εκεί στην ψηφοφορία θα προσπαθήσουμε λίγο να το, να το προσέξουμε αυτό και μετά, ε, ναι το είπα για την 9 αλλά και 76 με την 74 ε, δεν ε, δεν συνάδουν και στην 79 θα έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Ε, ελπίζω να μην έχουμε τέτοια, τέτοιες ε, περιπτώσεις ξανά. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Χάουταλα, να πω κι εγώ εξ αρχής ότι θέλω να εξηγήσω την ψήφο μου. Ε, ήταν ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό για τον εισηγητή, ειδικότερα λόγω του, των διακοπών του Πάσχα. Στη δική μας ομάδα υπάρχουν ε, ισχυρές ε, νομικές, ισχυρά νομικά επιχειρήματα σχετικά με αυτόν τον ε, μηχανισμό επίλυσης διαφορών για τις επενδύσεις και πραγματικά θέλουμε να δούμε πώς η γνωμοδότηση θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Αν τελικά αυτός λοιπόν ο μηχανισμός διαγραφεί από την γνωμοδότηση θα υπερψηφίσουμε, αλλιώς θα καταψηφίσουμε. Όμως είμαστε ανοιχτοί σε κάποιες διατυπώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ζητά ε, μία μελέτη βιωσιμότητα σε ένα μόνιμο ε, δικαστήριο, ε, αλλά θα θέλαμε γενικά έναν βελτιωμένο μηχανισμό. Ευχαριστώ. Thank you very much. We proceed to Σας ευχαριστώ. Περνάμε τότε στη ψηφοφορία. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τοπολογία 27 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ένα έλεγχο καλύτερα. Πολύ καλά. Και έχει εγκριθεί. 29. Με συγχωρείτε, 31 λέει ο Πρόεδρος. 31 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε ένα έλεγχο καλύτερα. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ένα έλεγχο εγκρίθηκε. Περνάμε στην 43. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Κάνουμε ένα έλεγχο. Δεν, ε, έχει, δεν μας φάνηκε έτσι από εδώ. Έχει εγκριθεί. Πάμε στη 42. Υπέρ. Κατά. Όχι, θα κάνουμε έλεγχο. Έλεγχο. Εγκρίνεται. Τοπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να κάνουμε ένα έλεγχο καλύτερα. Όλοι όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν έχουν ψηφίσει πέρα της ψηφοφορίας. Έχει εγκριθεί. Τεπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έχει εγκριθεί. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κάνουμε τον έλεγχο. Έχει εγκριθεί. Θα περάσουμε στο Με συγχωρείτε, έχουμε ένα ε, πρόβλημα με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Είμαστε στην τροπολογία 33. Υπέρ. ναι, είμαστε στην τροπολογία 33. Υπέρ. Εγκρίθηκε, ναι. Η 52 εγκρίθηκε, ναι. Και η 53 εγκρίθηκαν. Είμαστε λοιπόν στην 33, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε την τροπολογία 33. Έχει εγκριθεί. 97. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εξήντα δύο. Είμαστε τώρα στην τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλω να γίνει έλεγχος. Ελέγχουμε λοιπόν. 62. Έχει απορριφθεί σαφώς. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται κατά την άποψή μου, αλλά ας το ελέξουμε καλύτερα. Όντως έχει απορριφθεί. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε και αυτό. Ελέγχουμε την 65. Ε, Έχει εγκριθεί. Τροπολογία υπαριθμών 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έτοιμα για έλεγχο. Ελέγχουμε την τροπολογία 70. Έχει απορριφθεί. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Εκτός μικροφώνου. Ας... Ε, λέω ότι η 74 δεν, είναι, δεν συμφωνεί με την 76. Δεν είναι συμβατή. Όχι. Με συγχωρείτε να το ξαναπώ. Εκτός μικροφώνου έχουν λεχθεί. Ας ψηφίσουμε την τροπολογία 74. Πρώτα την 74, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Απορρίφθηκε. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Την βλέπω ως απορριφθήσα, αλλά ας κάνουμε ένα έλεγχο. Τοπολογία 72. Ναι, πράγματι έχει απορριφθεί. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας την ελέγξουμε. 76 λοιπόν, έλεγχος. Πραγματικά απορρίφθηκε. 73 υπέρ. Κατά. Απόχες. Νομίζω έχει εγκριθεί. Εγκρίν, εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Με συγχωρείτε, 78 διορθώνει ο Πρόεδρος. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Την 81 ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Στην λίστα ψηφοφοριών έχετε εδώ ε, τη χωριστή ε, ψηφοφορία μέχρι το Until Incorporated TTIP και το δεύτερο τμήμα από το SUD μέχρι το τέλος. Ε, υπάρχει αίτηση για χωριστή ψηφοφορία. Ναι, η 79 έχει καταπέσει, αν μιλάμε για την ίδια τροπολογία. Είμαστε στην 79, έτσι. Αυτή έχει καταπέσει. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε στην 82, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Με συγχωρείτε, έχει εγκριθεί. 83. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος παρακαλώ. Ελέγχουμε την τροπολογία 94. Εγκρίνεται. 90... 96. Τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά. Κάνουμε ένα έλεγχο. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος της τροπολογίας 98. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά ας το ελέγξουμε καλύτερα απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την 109. Ας ελέγξουμε την 109. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να αλλάξω τα γυαλιά μου μάλλον. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος. εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε εγκρίνεται 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά ας κάνουμε έναν έλεγχο. Εγκρίθηκε. 115 115 Υπέ Κατά Αποχές Απορρίπτεται Θέλετε να το ελέγξουμε Ωραία 115 και έχει απορριφθεί. 116 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Θέλετε να την αλλάξουμε. Όχι. Περνάμε στην τοπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. με συγχωρείτε, εγκρίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ελέγχου. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίθηκε. Ανθρωπολογία 7 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα καλύτερα να το ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριπτέται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τοπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Α, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. 16 μάλλον 15. Τροπολογία 15 φαίνεται να είναι συμβατή με τη 13. Άρα θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Ωραία. 15 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Και εγκρίθηκε. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 23 Είναι κανείς άλλος που επιθυμεί να ψηφίσει. Ωραία, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε επί του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Και έχει εγκριθεί. συγχωρείτε. Εικοσπέντε μέλη έχουν ψηφίσει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχει εγκριθεί λοιπόν. Συγχαρητήρια στον κύριο Φως. Θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου από αυτή την έκθεση. Wurde das registriert oder nicht? Ο εισηγητής δεν θέλει το όνομά του να αναγράφεται ως ε, το όνομα του εισηγητή. Κυρία Ρέγνερ, ο κύριος Κάστα θέλουν και αυτοί τα ονόματά τους να διαγραφούν, άρα θα παραμείνει χωρίς όνομα. και ο κύριος ε, Κώστα ως ε, ισχυώδης εισηγητής ε, θα ήθελε να αποσύρει το όνομά του. Thank Ευχαριστώ πολύ. Uh, silence in the hall. Παρακαλώ, ησυχία στην αίθουσα. Θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Ζαν Μαρί Καβαντά να αναλάβει την Προεδρία αυτής της Επιτροπής γιατί πρέπει να αναλάβω κάποια άλλα καθήκοντα. Ευχαριστώ τον κύριο Καβαντά.